Il Presidente. La seduta è aperta. Άρχεται η συνεδρίαση. οι αρμόδιες αρχές του Βασιλείου της Ισπανίας διαβίβασαν στον Πρόεδρο την εκλογή